της 22ης Μαρτίου του 2017 ε, έκανε παλήθευση των εξουσιών του κυρίου Αντ Κοντ και αποφάσισε να επικυρώσει την εντολή του, ε, τη θητεία του από τις 24 Φεβρουαρίου 2017.